Uh, Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Η Λίντα έχει αρχίσει, αργήσει λίγο, αλλά έχουμε με παρημένη μερίσια διάταξη. Συμφωνήσαμε λοιπόν με την ε, γραμματεία να ξεκινήσω εγώ τη συνεδρίαση μέχρι να έρθει η Λίντα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, η οποία είναι διαθέσιμη στους φακέλους σας. Συμφωνείτε. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Λόγω απρόβλεπτων απουσιών δεν έχουμε διερμηνία από τα κροατικά, υπάρχει όμως παθητική διερμηνία προς τα κροατικά. Όπως γνωρίζετε, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε τις Ευρωπαϊκές Μέρες Ανάπτυξης, το Τούρε Ταξί. Έχουν εγγραφεί περίπου 5.000 άτομα, που σημαίνει ότι θα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση που είχαμε ποτέ, εμβληματική πρωτοβουλία για το 2015. Ο πρόεδρος ε, Σούλτς ε, θα προλογίσει και θα έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας και του Λουξεμβούργου που θα παρίστανται και πολλούς ε, υψηλούς προσκεκλημένους. Θα συμμετέχουν έχουν και ευρωβουλευτές στις συζητήσεις στα διάφορα πάνελ Υπάρχει και ένα πάνελ το οποίο έχει οργανώσει η Επιτροπή μας την 5η το πρωί στις 9.45, 10 παρατέταρτο στο α2 ε, auditorium για το θέμα του πώς μπορεί η κατάλληλη συνεργασία να καταπολεμήσει την ε, ε, διαφθορά θα συμμετέχουν διάφορες συνάδελφοι. Ο συνάδελφός μας θα συντονίσει τη συζήτηση. Εγώ θα συμμετέχω, θα συμμετέχει και η Λίντα ε, στο τελευταίο πάνελ. Οι συζητήσεις ε, θα ε, μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου. Τις 2.30 την Πέμπτη θα γίνει μια κοινή συνεδρίαση ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ συντονιστών που θα είναι ανοιχτή ε, σε όλους τους συντονιστές για να συζητηθούν οι προτεραιότητες της 29ης ε, ε, Γενικής Συνάλευσης μαζί με τον κύριο Χάμπα Άσαντ και επίσης στις 6 ώρα θα ανοίξει μια προσωρινή έκθεση του Παρλαμεντάριου με φωτογραφικό υλικό για το θέμα των οικογενειακών γευμάτων, αυτά τα οποία μας φέρνουν όλους κοντά. Ξέρετε ότι ε, αρχές Μαρτίου ε, έγινε η έναρξη, η παρουσίαση των φωτογραφιών αυτών στο Κοινοβούλιο και το Παρταμεντάριουμ θα διαθέσει φυσικά τις φωτογραφίες και έτσι θα μπορούν να τις δουν πολλοί άλλοι ε, πολίτες. Θα υπάρξει και μια έκτακτη συνεδρίαση 9 με 12.30 την ε, ε, Πέμπτη το πρωί για, ε, μεταξύ ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ για να συζητηθεί το θέμα του Ιράκ. Θα συμμετέχει και ο Επίτροπος Τηλιανίδης και η κυρία Καν που είναι Γενικός Γραμματέας για θέματα ε, βοήθειας προς πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, τη Δευτέρα στις 6 Ιουνίου στο Στρασβούργο γύρω στις 7.45 το απόγευμα θα γίνει μια κοινή συνεδρίαση ΔΕΒΕ με την Επιτροπή Προϋπολογισμών, Ελέγχου συγγνώμη, του Προϋπολογισμού, όπου θα παρουσιαστεί η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ε, αξιολόγηση και το σύστημα παρακολούθησης ε, με βάση τα αποτελέσματα. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις της ε, Προέδρου Λίντα Μακάβαν, όπως τις διάβασα εγώ. Άρα τελειώσαμε και με τις ανακοινώσεις Προέδρου. Επόμενο σημείο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 20 Απριλίου 2015, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής της 20 Απριλίου είναι στο φάκελό σας. Αν έχετε παρατηρήσεις επί των πρακτικών, μπορείτε να ενημερώσετε τη γραμματεία πριν από το πέρας της συνεδρίασης. Εάν δεν λάβουμε παρατηρήσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο υπαριθμών 4 στην ημερήσια διάταξη τώρα. Έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών. Θα έχετε λάβει το σχέδιο αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών της συνεδρίασης ε, της 20ης Μαΐου του 2015. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις, παρακαλώ ενημερώστε τη γραμματεία μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. Αν δεν λάβουμε παρατηρήσεις, τότε θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και ε, οι αποφάσεις και οι συστάσεις των συντονιστών. Τώρα, ανακοινώσεις της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κάτι να μας ανακοινώσει. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε και αυτό λοιπόν το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 6. Ο ρόλος των τοπικών αρχών σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Έχουμε την εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ελένη Θεοχάρους. Please. Thank you, Chair. Well, uh, since I επειδή έρχομαι από μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ήμουν αναγκασμένη να ταξιδεύω όλη τη νύχτα για να είμαι εδώ, στην ώρα μου, Ελπίζω λοιπόν να έχετε το φάκελο, την έκθεση στο φάκελό σας και θα παρουσιάσω την έκθεση αυτή σχετικά γρήγορα, δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, προτιμώ να ακούσω τα σχόλιά σας. Η επικεφαλίδα είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Αυτό είναι ο τίτλος της έκθεσής μου και εγώ ανέλαβα να συντάξω αυτή τη σημαντική έκθεση για το σημαντικό θέμα με στόχο να αναγνωριστεί η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο επίσης να υπάρχει στρατηγική για να βελτιωθούν, ε, βελτιωθεί η απόδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης για να πετύχουμε το στόχο μας που είναι να υπάρχουν ευημερούσες ε, κοινωνίες στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Με αυτή τη στρατηγική ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αναπτυξιακά προγράμματα με ένα πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η σημασία του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα προφανώς και σε μια σειρά ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και σε άλλες πολλαπλές προσεγγίσεις στις οποίες έχει προβεί, έχουν προβεί τα Ηνωμένα Έθνη. Συμφωνώ μαζί τους με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη και αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσής μου. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρει προστιθέμενη αξία ε, στη διαδικασία της ανάπτυξης, μειώνοντας τις προσπάθειες, ε, μειώνοντας τη φτώχεια, συντονίζοντας και στηρίζοντας ε, άλλες ΜΚΟ και βελτιώνοντας την κυβερνητική διαχείριση. Ξέχασα να ευχαριστώ τους αδέλφους μου που με βοήθησαν να συντάξω την εκθεσή μου. Το θυμήθηκα τώρα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι ο ρόλος τοπικής αυτοδιοίκησης ε, ε, ε, στο έργο των ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων της ε, χιλιετίας. Σημαντική, σημαντικά είναι έργα υποδομής, όπως επίσης και η διάδοση των πρωτοβουλειών ε, συντονισμού Αναφέρομαι επίσης ε, στη διαδικασία μετά το 2015, προβάλλοντας κυρίως την ανάγκη να υπάρχει ένα σαφές όραμα για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων ε, της συνάντησης του Ρίου και εκεί υπογραμμίζεται ο ρόλος της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζω ότι θα πρέπει οι πόλεις να έχουν μια αυτονομία. Έτσι λοιπόν καθίζεται σαφε ότι πρέπει να υπάρχει μια οικουμενική συνεργασία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η εκπρόσωποι τους θα μπορούν να συνεργάζονται για να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην κοινή γνώμη και να αναλαμβάνονται περισσότερες πρωτοβουλίες. Κατόπιν εστιάζουμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι ένα σημαντικός παράγον για να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μέσα από ΣΔΙΤ να ε, εφαρμόζουν μηχανισμούς αποτελεσματικής λογοδοσίας και να ορίζουν ε, ρήτρες για το περιβάλλον. Οι συνεργασίες και οι μηχανισμοί που έχουν καθοριστεί για να υπάρχει διάλογος ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία των πολιτών και αυτοί οι μηχανισμοί είναι πολύ χρήσιμοι. Η υποστήριξη λοιπόν ε, της λογοδοσίας είναι άλλο σημαντικό θέμα γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να λογοδοτούν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς άμεσα ενδιαφέρον με ε, διαφάνεια να ενισχύεται η συμμετοχή των γηγενών, ε, των μειονοτήτων, των προσφύγων στις αναπτυξιακές στρατηγικές και στον προγραμματισμό των επενδύσεων. Ένα άλλο θέμα το οποίο απορρέει από τη δική μου την εμπειρία είναι ότι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική σημασία. Ε, να εφαρμόζονται πολιτικέ προ όφελο τη κοινωνία για χρηστή διακυβέρνηση και να υπάρχει αγώνα κατά τη διαφθορά αλλά και τη γραφειοκρατία. Επίση, είναι ένα τρόπο για να ελέγχει κανεί ε, την παρανομία, το ξέπλυμα ε, χρήματος και να υπάρχουν ίσοι όροι στη φορολογία. Μία άλλη σημαντική πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι η ενίσχυση στην κινητοποίηση των πόρων, να υπάρχουν συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε και επανένταξη του, ε, του, του, κρατικού τομέα χωρίς να αποταρρύνεται το ιδιωτικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αφέμαξη εγκεφάλων, να βελτιώνεται προφανώς η βημερή αυτό το θέμα το έχουμε ε, τονίσει επανειλημμένα κυρίως σε σχέση με την εξάλληψη της φτώχειας, αν θυμάται. Έτσι λοιπόν η άμεση εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή ε, στην αναπτυξιακή πολιτική είναι μία δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν κρίσει. Με αυτή μου την έκθεση προσπαθώ να αντιμετωπίσω το υπάρχον πλαίσιο και να δώσω τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσουν ω παράγοντε τη ανάπτυξη σε συμφωνία με τι γενικέ αρχέ ε, που υπάρχουν σε διεθνέ επίπεδο και παράλληλα θέλω να υπάρχει νομική συνέπεια όσον αφορά τις αρμοδιότητες και την ευθύνη που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα περιφερειακός, τοπικός τομέας θα πρέπει να εκπροσωπείται καλύτερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να εισακούται και η φωνή του σε, σε ομάδες διεθνών δωρητών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ειδικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στην τοπική αυτοδιοίκηση να συντονίζει καλύτερα τις ενέργειές της, καλύτερο συντονισμό με ως χαρά στην ευρωπαϊκή πολιτική, βελτίωση της συνεργασία ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις δωρήτριες χώρες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο προσθέτει στην έκθεση. Έτσι λοιπόν η ανταλλαγή προγραμμάτων βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση Ευρωπαϊκή Ένωση και την τοπική αυτοδιοίκηση των αναπτυσσομένων χωρών ή ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο είναι καθοριστική σημασία. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν υπάρχει ένα σημαντικό πρόγραμμα για μια συγκεκριμένη περιοχή μπορούμε ε, να στέλνουμε εκπροσώπους τοπική αυτοδιοίκησης από μια άλλη περιοχή και με τον τρόπο αυτό προκύπτει πολλαπλασιασμό, στοιχείο πολλαπλασιασμού ε, με βάση μια έκθεση. Αυτή λοιπόν η έκθεσή μου και περιμένω τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε την κυρία Σιγήτρια. Το επώνυμό σας είναι σχεδόν δύσκολο σαν το δικό μου να το προφέρει κανείς. Ναι, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το επώνυμό μου, είναι η χάρη του Θεού. Εγώ είμαι από τη Λαπωνία, από τα πιο βόρεια μέλη δηλαδή του Κοινοβουλίου, εσείς από τα πιο νότια. Ωραία, τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κύριος Μανσκούρ, από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε στο μέσο μιας εξαιρετικής χρονιάς για την βιώσιμη ανάπτυξη η έκθεση δείχνει πόσο ο ρόλος των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών ε, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και να ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ποιότητα του έργου της και την ε, συνέπεια και τον πλούτο των σκέψεών της επί του ζητήματος. Η ευθύνη των ε, κρατών είναι ένα προφανές στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε την... το έλλειμμα ανάπτυξης, όμως πρέπει να εξετάσουμε και άλλα στοιχεία, όπως τα επεσήμανε η συγγήτρια. Εγώ βρέθηκα ε, επικεφαλής μιας κοινότητας ε, για πάνω από έξι χρόνια και συμμετείχα σε πολλά τέτοια προγράμματα στην Καραϊβική και μπορώ να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι έχει ανεκτήμητη προστιθεμένη αξία αυτό το έργο των ανταλλαγών μεταξύ τοπικών ε, αρχών. Γι' αυτό και αυτή η έκθεση, κατά τη γνώμη μου, είναι μία πολύτιμη ευκαιρία να απευθύνουμε έκκληση, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ε, και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, να έχουν ε, μία πολυεπίπεδη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Το σχέδιο έκθεσης Δείχνει λοιπόν ξεκάθαρα γιατί οι τοπικές αρχές θα αποτελέσουν και είμαι ένα πολύτιμο εργαλείο για να εξαλείψουμε τη φτώχεια, να προωθήσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση, να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής. Ο παγκόσμιος πληθυσμός ε, αστικοποιείται όλο ένα και περισσότερο. Και τα δημογραφικά στοιχεία και προγνωστικά για τα επόμενα χρόνια μας δείχνουν ότι αυτή η τάση θα ενταθεί, ιδίως ε, στις ε, υπαναπτυξή χώρες. Βασικές υπηρεσίες όπως η παιδεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η πρόσβαση στο νερό ε, και το καθεξής. Σε αυτά τα σημεία λοιπόν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο όπως εντάσσεται και στο πλαίσιο ε, των ε, στόχων για τη χιλιετία αλλά και για των στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι τοπικές αρχές είναι αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα των του κόσμου, των πολιτών. Γι' αυτό και ε, συνιστούν ένα δίκτυο ε, δημοκρατικού βίου και έτσι και ο κάθε πολίτης μπορεί να συμμετάσχει στο δημοσιοβίο. Οι πρόσφατες καταστροφές μας έχουν δείξει και την ε, απίστευτη αλληλεγγύη που μπορεί να δείξει ο άνθρωπος όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Τα ε, ταμεία αλληλεγγύης των ΗΠΑ, της Γαλλίας για να βοηθηθούν τα θύματα και οι επιζώντες ε, ε, του σεισμού στο Νεπάλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι πολύ απλό. Οι τοπικές αρχές θεωρούνται θεωρείτε ότι βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων και στηρίζονται και με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση είναι πως όχι, δεν στηρίζονται επαρκώς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συμβολή, η μας προς την εξωτερική πολιτική επιβεβαιώθηκε από τα όσα υιοθετήθηκαν το 2005 και μετά επανεβεβαιώθηκαν από τα έργα της Επιτροπής το 2018 και 2013 και από την έκθεση του Κοινοβουλίου το 2007 και το 2013. Σε διεθνές επίπεδο, οι στόχοι για τη χιλιετία βρίσκονται στην ε, πρώτη γραμμή, συγγνώμη, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν ε, συμβάλει συστηματικά και αποφασιστικά στην ομάδα εργασίας ε, του ΟΗΕ για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η έκθεση είναι επίσης μια ευκαιρία να ε, κάνουμε ορισμένες προτάσεις για το μέλλον. Σε ό,τι φορά αρχικά την χρηματική υποστήριξη. Το πλαίσιο που υπάρχει από το 2007 έχει αποδείξει το ρόλο του, αλλά πλέον δεν επαρκεί. Γιατί είναι πολλές οι προκλήσεις από την ε, αποκέντρωση στις χώρες εταίρους. Πρέπει να αποτελέσει λοιπόν αυτό ένα τομέα συγκέντρωσης των χρηματικών πόρων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Μιλάμε για την ε, διάρκεια και την αποτελεσματικότητα των ε, προγραμμάτων αποκέντρωσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες εταίρους. Η ΟΤΑ, εξάλλου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε άλλες καινοτόμε πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί που δεν εντάσσονται στις ιδιαιτερότητες ε, των τοπικών αρχών ε, των χώρων εταίρων. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την συστηματική συμπερίληψη των ΟΤΑ, σε ό,τι αφορά τον ε, πολιτικό διάλογο στις ε, χώρες εταίρους. Οι τοπικές αρχές και οι ενώσεις ε, εκεί δεν γνωρίζουν ακόμα αρκετά την πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν γνωρίζουν ούτε πώς ούτε γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν στις αντιπροσωπείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 84 από αυτές τις οργανώσεις ζήτησαν χρηματοδότηση από το ε, θεματικό πρόγραμμα το σχετικό για να συνεργαστούν με τοπικές αρχές. Αυτή η εξέλιξη θεωρώ ότι είναι θετική. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Γι' αυτό προτείνω να υπάρχει ε, εκπρόσωπος τοπικών αρχών ε, σε κάθε χώρα αναπτυσσόμενη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω προτάσεις, κυρία Συγήτρια, προτάσεις τροπολογιών, για να εμπλουτίσουμε ακόμα παραπέρα το εξαιρετικό αυτό κείμενο. Σας ευχαριστώ. you. And, um, thank, I Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Βάιρεν που ανέλαβε ε, το Προεδρείο. Το Eurostar δεν είχε τρένα σήμερα και χρειάστηκε να έρθει ο αεροπορικός, γι' αυτό καθυστέρησα. Ο λόγος στην κυρία Μπεατρίς Μπεθέρα τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι από πλευράς φιλελευθέρων δύο σχόλια θα θέλαμε να κάνουμε για την έκθεση αυτή. Ο στόχος της έκθεσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στο να καθορίσουμε τον σημαντικό ρόλο των ε, τοπικών αρχών ε, για την ε, ένταξη των διαστάσεων της ανάπτυξης. Ε, εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και προς αυτό θα συνεισφέρουμε να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Και γι' αυτό και ο συνάδελφος Μπέρενς και εγώ ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για προκειμένου να καθορίσουμε ποιος είναι ο χώρος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουν να δράσουν άμεσα σε τοπικό επίπεδο ε, μήπως θα πρέπει να γίνει μέσω διαμεσολάβησης και πάλι των εθνικών αρχών. Αυτή η δράση να μπορούμε να δρούμε άμεσα χωρίς διαμεσολαβικές θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε ποιες πτυχές ε, ε, θα πρέπει να τελειοποιήσουμε σε μια τέτοια έκθεση, κυρίως σε τρεις πτυχές οι οποίες κατά την άποψή μας είναι κλειδί. Καταρχάς ε, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι τοπικοί φορείς να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, την τεχνολογία, την αξιολόγηση και τις δυνατότητες εν γέννη να δράσουν φτάσουν σε τοπικό επίπεδο και να αναπτύξουν τις πολιτικές τους και σε κοινωνικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να συνεισφέρουν και επίσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για μια έκθεση που πρέπει να είναι τόσο συγκεκριμένη όπως η έκθεσή σας να ε, σταθούμε και στα θέματα φύλου ε, οριζόντια σε όλες τις πτυχές, να μην υπάρχει απλώς μια αναφορά που λέει ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε ε, για τους στόχους της χιλιετίας και τη διάσταση των φύλων, αλλά να υπάρχει η ίδια η έννοια της συμμετοχής. Οι τοπικές αρχές προκειμένου να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ε, ε, ισότητα των φύλων, θα πρέπει ε, ίσως να ενημερωθούν από γυναίκες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο πολιτικό βίο. Το να δράσουμε λοιπόν αποτελεσματικά και ως ψηφοφόροι αλλά και ως εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φυσικά όταν υπάρχει κατάλληλη ισορροπία που θα σε επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται και να εφαρμόζεται αυτή η ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές. Και τέλος να αναφερθώ και σε κάτι που αναφέρεται για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη είναι αυτό, όχι μόνο για να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά τους ως προς τις γνώσεις και τη δυνατότητα που έχουν για να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, αλλά και κατά την εκτέλεση. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν αρκετοί αυτόχθονες πληθυσμοί όταν ε, ε, περάσαμε στη διαδικασία εκτέλεσης των ε, προγραμμάτων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και αυτή τη δυνατότητα και να μην τους λαμβάνουμε υπόψη μόνο εκ των πρετέρων, αλλά και εκ των υστέρων κατά την εκτέλεση των διαφόρων θεμάτων. Συνοψίζοντας λοιπόν, ως ε, προτεραιότητα θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να μας επιτρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι, κυρίως όσον αφορά τον αρχικό ε, ορισμό, πού ακριβώς δρούμε, ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής δράσης μας ε, και την άμεση σχέση μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τοπικού ε, ε, τοπικής αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ η Μαρία Χόιμπουκ από πλευρά πρασίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την καλή τη έκθεση που περιλαμβάνει πολλά σημαντικά θέματα. Πράγματι χρειαζόμαστε ενίσχυση για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και είναι σημαντικό ε, να παίξουν σε αυτή την προσπάθεια πολλοί παράγοντες ε, το δικό τους το ρόλο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μία πρόκληση το να προσφέρουμε αποτελεσματική βοήθεια, διότι ο συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους φορείς δυστυχώς λείπει και αυτό λείπει και από την έκθεση. Δηλαδή αν δεν υπάρχει συντονισμός των διαφόρων φορέων, χωρίς συντονισμό δεν μπορεί να προσφερθεί αποτελεσματική βοήθεια. Αυτό πρέπει να προσθεθεί στην έκθεση, γιατί σε επίπεδο ορχής ε, πρέπει να τηρούνται οι στόχοι της αποτελεσματικότητας. Έτσι λοιπόν, όταν σε αναπτυσσόμενες χώρες δραστηριοποιούνται φορείς, είναι απαραίτητο η δραστηριότητά τους να περιλαμβάνεται σε όλα τα εθνικά προγράμματα. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να επιτύχει έχει τη συνέπεια σε όλα τα επίπεδα. Συντονισμός λοιπόν. Ο συντονισμός, επαναλαμβάνω, των φορέων λύπη πρέπει να προσθεθεί στην έκθεση. Και εκείνο το οποίο επίσης είναι απαραίτητο είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η υποχρέωση για λογοδοσία. Γιατί μόνο αν υπάρχει υποχρέωση για λογοδοσία ε, μπορεί πράγματι κανείς να επιτύχει τους στόχους του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πολύ για την έκθεσή σας και εμείς ως πράσινοι θα καταθέσουμε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει σε αυτή την έκθεση και συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των υπολείπων συναδέλφων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση δεδομένου, δεδομένων των ιστορικών εξελίξεων που περιμένουμε αυτή τη χρονιά. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας ως ε, μία κίνηση ε, προς ε, τις εξελίξεις και τις επιτυχίες που θέλουμε να πετύχουμε. Είναι ιστορικός ο ρόλος των τοπικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν μεταξύ κρατών μελών, όμως ε, έχουμε πλούσια παράδοση από τις ε, τοπικές αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πήρα το λόγο για να κάνω τις εξής παρατηρήσεις μόνο. Αρχικά, στη δική μου εκλογική περιφέρεια στην ε, Ιρλανδία, ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές Ιρλανδικές τοπικές αρχές έχουν συνάψει πολύ σημαντικές σχέσεις, εταιρικές σχέσεις με άλλε τοπικέ αρχές σε άλλα μέρη του κόσμου. Κυρίως ε, για την κατάρτιση, την οικονόμηση του δυναμικού και το καθεξής. Εξαιτία αυτή ακριβώ ε, τη ιστορική γνώση και τη οικοδόμηση ε, δυνατοτήτων, οι τοπικέ αρχέ στην Ευρώπη μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα για να συνάψουν τέτοιες εταιρικέ σχέσεις με χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου όχι μόνο για την καλύτερη χωροταξία, για, την, για περιβαλλοντικούς λόγους, καλύτερες διαβουλεύσεις για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους λοιπόν για να ενθαρρύνουμε περισσότερες τοπικές αρχές να αναλάβουν αυτό το ρόλο που θέλουμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων στις αναπτυξιακές μας προτεραιότητες, τότε πρέπει οι τοπικές αρχές να έχουν αποτέλεσμα και αντίκτυπο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Να τους δίνουν δηλαδή τις ικανότητες να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά και να χαρτογραφούν ζητήματα, όπως επεσήμανε πολύ σωστά η συγγήτρια, είτε στο ζήτημα της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, στον τομέα που εγώ ο ίδιος εξέτασα τον περασμένο μήνα με τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα και τι ρόλο παίζουν εκεί οι ε, τοπικές αρχές, πώς γίνεται κανονικά αυτός ο διάλογος με τις τοπικές αρχές στα, στις χώρες των προγραμμάτων και στις συμφωνίες που συνάπτουμε. Βρισκόμαστε ήδη δηλαδή σε επαφή με τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης για να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε τα, τα, τους στόχους μας. Πολλές είναι οι δυνατότητες εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια που τα έθιξε όλα αυτά, γιατί αυτή τη χρονιά που ελπίζουμε να έχουμε μια ιστορική συμφωνία, πρέπει πραγματικά να τονίσουμε τον ρόλο της τοπική αυτοδιοίκησης και τον ε, τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε τους ε, στόχου που θέλουμε όλοι ω Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Νόμπετ Νόιζα. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω ακριβώς εκεί που σταμάτησε ο κύριος Χέις, ο οποίος ε, αναφερθήκε στο ρόλο της, των τοπικών αρχών στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει αυτό να το αναφέρουμε στην έκθεση. Υπάρχουν ε, πολλές αδελφοποιήσεις ε, ανάμεσα σε πόλεις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και αδελφοποιήσεις ανάμεσα σε περιφέρειες που αυτές λειτουργούν θαυμάσια. Ε, και χωρίς βοήθεια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο στην Επιτροπή των Περιφερειών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ε, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφέτος, κυρίως ε, στο πλαίσιο της ε, ανάπτυξης. Εγώ προέρχομαι από τη Ρινανία Παλατινάτο. Ε, τέσσερα εκατομμύρια είναι το κρατήδιό μας. Συνεργαζόμαστε με τη Ρουάντα και υπάρχουν περίπου 200 αδελφοποιήσεις και αυτές ακριβώς βοηθούν στο να υπάρχει ευαισθητοποίηση στην δική μας την κοινή γνώμη. Αυτή η ευαισθητοποίηση είναι κάτι το οποίο οποίο νομίζω μπορείτε να το προβάλλετε στην έκθεσή σας. Πέρα από αυτό το θέμα της ευαισθητοποίησης, νομίζω όλα τα άλλα ε, τα έχετε αναφέρει. Θαυμάσια παρουσιάζεται τη σημασία των τοπικών αρχών, μόνο που νομίζω ότι και εμείς ε, στην Ευρώπη πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πράγματι όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν έχει στήσει κάποιος άλλος το λόγο. Από την Επιτροπή όμω, Μισελ Λελός, έχετε ζητήσει το λόγο από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Την περασμένη εβδομάδα να αναφέρω ότι στην ομάδα των σοσιαλιστών ακούσαμε σε ένα σεμινάριο τι συνδέσεις μεταξύ σχολείων στον Ρενό Βασίλειο και ε, προσφύγων σύρων. Υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε λοιπόν τώρα ανάπτυξη τέτοιων δεσμών μέσω ακριβώς τοπική αυτοδιοίκηση. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Λαλό. Ευχαριστώ. Αρχικά, εν είδη εισαγωγή, θα θέλω να πω ότι οι συστάσει και τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση συνάδουν απολύτω με την πολιτική, ιδίω ε, τη τελευταία ανακοίνωση του 2013, που αναφέρονται τέσσερι προτεραιότητε. Αποκέντρωση, αύξηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αστικοποίηση, βιώσιμη βεβαίω. Και το τέταρτο σημείο, το οποίο κατά γνώμη δεν έχει υπογραμμιστεί αρκετά, είναι ο ρόλος της ε, ε, τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό, περιφερειακό ή και παγκόσμιο επίπεδο. Κατανοούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τοπικών Αρχών είχε αποφασιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και μεταξύ άλλων ο στόχος παριθμών 11 που αφορά ακριβώς την αστικοποίηση είναι κάτι το οποίο στηρίχθηκε από τις τοπικές αρχές. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση υπενθυμίζει όλα τα εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα στοιχεία για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή βοήθεια. Από την άλλη θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι ίσως κάτι ξέφυγε από την εισηγήτρια. Αυτό που μιλάμε εδαφική προσέγγιση. Είναι μία μέθοδος, εντάξει όχι ακριβώς μέθοδος, αλλά ένας τρόπος ανάπτυξης της επικράτειας, όπου θέτουμε τέσσερα στοιχεία της ανάπτυξης. Έχουμε το κράτος βεβαίως, με πολύ κεντρικό ρόλο, τον ιδιωτικό τομέα, αναφέρεται αυτό, κοινωνία των πολιτών με όλη την πολυμορφία της, ε, ΜΚΙΟ, ε, συνδικαλιστικέ ενώσει και, άλλες, ε, και άλλοι οργανισμοί. Και σήμερα μιλούμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικέ αρχέ. Θα ήταν καλό να λάβουμε υπόψη και αυτό το στοιχείο που επιχειρεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τον προγραμματισμό υπάρχει μια θεματική που έχει ήδη υπογραμμιστεί. 84 χώρες ακριβώς ε, ακολουθούν την προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που θα υποφεληθούν μέσα στα επόμενα χρόνια ε, τέτοιων ευρωπαϊκών πόρων. Μετά έχουμε και εθνικές αρχές των χωρών εταίρων και το σημείο στήριξής μας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη. Έτσι προσεγγίζουμε εμείς αυτή τη θεματική. τα όσα αναφέρονται για την αποκέντρωση. Υπάρχουν πολλές ε, ε, χώρες ε, σε διμερές επίπεδο που εργάζονται με τις τοπικές αρχές για την αποκέντρωση, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική ανάπτυξη. Και άλλες δράσεις βεβαίως για την οικοδόμηση επιχειρησιακών ικανοτήτων των τοπικών αρχών. Αυτά είχα να πω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή έκθεση. Αναφέρθηκε από πολλούς ε, προ... Βρισκόμαστε σε μια κέρια χρονική στιγμή και είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι αρχές ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ως ε, βασικός παράγοντας. Αυτό κάνουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ να ληφθεί και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θεοχάρου θέλει το λόγο και πάλι. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους συναδέλφους και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά τους. Θα τα λάβω σοβαρά υπόψη μου και φυσικά προσβλέπω στην αγαπητή συνεργασία με τους κύριους ηγητές προκειμένου να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική έκθεση εν τέλει. Το μόνο σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι ότι στις περισσότερες από τις κοινότητες της υποσαχάριας Αφρικής η ισότητα των φέλων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που βιώνουμε εμείς στην Ευρώπη. Σας διαβεβαιώ. Thank you. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στις 23 Ιουνίου. Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο σημείο 7, πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου Και έχουμε και το 8 που είναι δύο αντίστοιχα πράγματα, δύο γνωμοδοτήσεις για την τροποποίηση της συμφωνίας ε, του Μαρακές, του πρωτοκόλλου για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Χρειάζεται ε, σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και χρειαζόμαστε δύο εκθέσει. Η μία θα λέει κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί σύμφωνη γνώμη και ο εισηγητή ε, προτείνει ε, να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα. Και η δεύτερη, επειδή η επί αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή ΙΝΤΑ ετοιμάζει ένα ψήφισμα το οποίο θα συνοδεύει το κείμενο, μπορούμε να συνεισφέρουμε και στο ψήφισμά του. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε δύο διαφορετικέ νομοδοτήσει. Η μία απαντά καταφατικά ή αρνητικά και η άλλη είναι ε, τροπολογίες ε, στο ψήφισμα της Επιτροπής ε, ΙΝΤΑ για την Συμφωνία Διευκόλυνση Εμπορίου. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης, ο Ντόρου Κλάντιαν Φρουντζουλίκα, δεν είναι εδώ σήμερα. Θα μιλήσει εκ μέρους του κυρίου Σνόιζε και θα παρουσιάσει την έκθεσή του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω τις απόψεις του συναδέλφου για τη νέα τροποποίηση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Η συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία συμφωνήθηκε στις, ε, το Δεκέμβριο του 2013, ε, είναι ουσιαστικά το ε, βασικό αποτέλεσμα του γύρου της Ντόχα. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη ροή προϊόντων μέσω απλούστευσης και εξυγχρονισμού, κυρίως ε, των τελωνιακών απαιτήσεων που ορισμένες φορές αποτελούν πρόσκομα για το εμπόριο. Από αναπτυξιακή σκοπιά η συμφωνία θα μπορούσε να θεωρηθεί ιστορική σημασίας επειδή υπάρχουν ε, ε, ευελιξίες χωρίς προηγούμενο για τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες μέλη του ΠΟΕ. Υπάρχει δυνατότητα να καθορίζουν μόνες τους πότε ε, θα εφαρμόζουν το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, για κάθε ένα από τα μέτρα που προβλέπεται. Η προσέγγιση αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη καινοτομία, διότι αποτελεί και ορόσημο για τις μελλοντικέ συμφωνίες. Οι εκτιμήσεις του ΟΣΑ είναι ότι η εφαρμογή όλων των μέτρων που προβλέπονται από τη Συμφωνία του ΠΟΕ μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος των εμπορικών συναλλαγών κατά 13-15% στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επομένως, αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή θα μειώσει το χρόνο και το κόστος του εμπορίου. Επίσης, θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις επιχειρήσεις τους, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενσωματωθούν καλύτερα στις ε, περιφερειακές και παγκόσμιες αξίες ε, ε, διανομής, αλυσίδες διανομής. Πρέπει βέβαια να ε, γίνει εφαρμογή της συμφωνίας, ε, να υπάρχουν 400 εκατομμύρια ευρώ ε, σε διάρκεια 5 ετών ως τμήμα του εμπορίου. Ο εισηγητής μας προτείνει να δώσουμε τη συμφωνή γνώμη μας για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας διευκόλυνσης εμπορίου και όσον αφορά τώρα τη γνωμοδότηση του μη νομοθετικού ψηφίσματος, θα προτείνει κάποιες τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, την περιφερειακή ολοκλήρωση, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ε, στοιχεία για την ανθρωπιστική βοήθεια και πώς μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως επιθυμεί κάποιο ε, συνάδελφο να λάβει το λόγο. Η κυρία Χόιμπρουκ, παρακαλώ. Τώρα, για τι πράγμα θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε μόνο για το ψήφισμα που μπορούμε να πούμε μόνο ναι ή όχι ή θα μιλήσουμε και για τη γνωμοδότηση όπου μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Δεν το έχω καταλάβει, μπορείτε να μου το διευκρινίσετε. Πρόεδρος, θα έπρεπε πράγματι να το έχω διευκρινίσει. Συζητάμε και για τα δύο. Δηλαδή, συζητάμε για το κατά πόσον θα συνενέσουμε σε αυτή την έκθεση ε, και επίσης συζητάμε και για το ψήφισμα. Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος για να αλλάξει, να τρόπο χρησιμοποιήσει κανείς ε, την πρώτη γνωμοδότηση είναι να πει ναι ή όχι. Το δεύτερο είναι, όπως σας είπα, ένα κανονικό ψήφισμα ε, και εκεί μπορεί κανείς να καταθέσει τροπολογίες. Άρα σχόλια και για τα δύο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και συγκεκριμένα. Η θέση των αναπτυσσομένων κρατών νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη. Ε, με βάση το αναπτυξιακό κέντρο που ασχολείται με αυτά τα θέματα υπάρχουν κάποια θέματα που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο και αυτά τα θέματα δυστυχώς δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη στην έκθεση. Καταρχήν οι ε, βιομηχανικές χώρες ε, θα επωφεληθούν περισσότερο από τις αναπτυσσόμενες χώρες διότι ε, από το ψήφισμα αυτό, αν εφαρμοστεί, θα μπορούν οι αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αναπτυσσόμενες και όχι τα νάπαλιν. Οι, οι εισαγωγές ε, για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες θα αυξηθούν και αυτό δεν θα επηρεάσει τις εξαγωγές τους. Περισσότερες εξαγωγές χωρίς εξαγωγές. Επίσης, στην έκθεση υπάρχουν κάποια στοιχεία που αφορούν τα κλωστοεφαντουργικά, κλωστοεφαντουργικά όμως σε σχέση με εισαγωγές και όχι εξαγωγές αναπτυσσομένων κρατών. Αύξηση των εισαγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό θα οδηγήσει ε, σε επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου των ε, αναπτυσσομένων κρατών, κάτι που αντιβαίνει αρχές του ΠΟΕ. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που δυστυχώς δεν αναφέρεται. Και κάτι άλλο, πρόκειται για το κόστος. Οι νέες διαδικασίες ε, σχετικά με τις ε, διασυνοριακές διεργασίες αυτά που καλούνται να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις πολύ συχνά συνδέονται με επιπρόσθετο κόστος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις αναπτυγμένες χώρες, γιατί οι τελευταίες ε, έχουν υιοθετήσει τις περισσότερες πρακτικές και ως εκ τούτου καλύπτονται οι δικές τους οι ανάγκες. Άρα δηλαδή υπάρχουν οι προδιαγραφές, γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι βέλτιστες πρακτικές, όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ακόμα αυτές τις προδιαγραφές. Άρα το λιγότερο που μπορούμε να ζητάμε είναι για τις αναπτυσσόμενες χώρες να προβλεφθεί ένα πλαίσιο, μια ευελιξία εφαρμογής ανάλογα με τις δυνατότητες δυνατότητές τους. Και επιπλέον οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρέπει να υποχρεωθούν να εισάγουν ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές εάν δεν είναι ε, σε θέση να μπορούν να τηρήσουν όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτό είναι το δεύτερο που δεν αναφέρεται στην έκθεση και το τρίτο αφορά στον ε, περιορισμό των δασμών, ε, των δασμολογικών και φορολογικών εσόδων. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, αν καταργηθούν οι δασμοί, αυτό σημαίνει για τις αναπτυσσόμενες και κυρίως για τις πολύ λίγο αναπτυγμένες χώρες ότι δεν θα έχουν κρατικά έσοδα γιατί στις χώρες αυτές τα περισσότερα έσοδα του κράτους προκύπτουν από τους δασμούς. Ούτε και αυτό το θέμα αναφέρεται στην έκθεση. Αυτές τις παρατηρήσεις είχα να κάνω και ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρονς έχει το λόγο. Ε, μία απλή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο βαθμό η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ επενεύει στις διαδικασίες ε, που εξετάζουμε εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Δεν έχει δει κανένα άλλο τον λόγο. Αλλά και εγώ να θέσω ένα ερώτημα προς την Επιτροπή. Κατόπιν των όσων είπε και η Μαρία Χόιμπρουκ. Η αιτιολόγηση του συγκεκριμένου αναφέρει ότι θα υπάρχει νέα προσέγγιση όπου οι αναπτυσσόμενε χώρες θα μπορούν να προσδιορίσουν οι ίδιες ε, την ταχύτητα εφαρμογής των διατάξεων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το όφελος ε, για τις χώρες αυτές της προσχώρηση τη αυτή τη συμφωνία, ό,τι αφορά τη δική γενική διεύθυνση. Και δεύτερον, αυτή η διάταξη για τον ΠΟΕ πώς συνδέεται με τον TTIP, άλλες διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και αναδυόμενων οικονομιών. Πώς όλα αυτά θεωρείτε ότι συνδυάζονται. Γκί Πλατών, δεν ξέρω πώς να το πω. Α, όχι. Αλμπέρ Λεβάντε τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Δεν ξέρω αν τα πάει καλά. Παρακαλώ, ενημερώστε μας. Να, Αλμπέρ Λεβάντ. Ευχαριστώ. Εντάξει, είναι περίεργο το όνομά μου, γκρικό. Πρώτα βάζουμε εμεί το επώνυμο, σαν τους Κινέζους. Θα απαντήσω, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι η έκθεση ήταν εξαιρετική. Α, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε. Και επειδή ακριβώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, δεν μπορώ να απαντήσω εξ ονόματο ε, τη ΔΕΦΚΟ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Και οι δύο αναφερθήκατε στο ζήτημα τη ειδική και προτιμησιακή ε, ε, μεταχείρισης ε, για τις αναπτυσσόμενες ε, και λιγότερο επιτυχημένες χώρες σε αυτή τη συμφωνία και πράγματι είναι ένα από τα πλέον καινοτόμα στοιχεία της συμφωνίας. Οι υποχρεώσεις μπορούν να ταξινομηθούν από τις χώρες αυτές σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η κατηγορία Α, οι υποχρεώσεις δηλαδή που οφείλουν να εφαρμόσουν άμα τη θέση ισχύει τη της Η κατηγορία Β δεσμεύσεις όπου χρειάζεται ένα επιπλέον μεταβατικό ε, στάδιο, μια περίοδος προσαρμογή και εφαρμογή και κατηγορία Γ που είναι και πλέον σημαντική και να θυμάστε ότι έχουν απόλυτη ελευθερία να ταξινομήσουν όπω θέλουν τις ε, δεσμεύσει αυτές όπου η εφαρμογή θα εξαρτάται από την δυνατότητα εφαρμογή. Και είναι κάτι το οποίο εγγράφεται ξεκάθαρα στην ε, συμφωνία. Οι δωρητές ε, ανέλαβαν την ε, δέσμευση να οικοδομήσουν ακριβώς και να βελτιώσουν αυτή τη δυνατότητα. Όλες... Το, το μόνο λοιπόν που πρέπει να κάνει η αναπτυσσόμενη χώρα ή η λιγότερο αναπτυγμένη χώρα είναι να επισημάνουν στον ΟΣΑ ότι αυτές οι δεσμεύσεις βρίσκονται στην κατηγορία Γ. Και από εκεί και πέρα ε, θα τεθούν ε, στο στόχο αυτές οι ανάγκες ακριβώς μέσω των 8 προγραμμάτων Μπορεί να είναι διμερή, να τα χειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, το Δουνουτού ή ο ίδιος ο ΩΣΑ και όταν η πτωσόμενη χώρα αποφασίσει ότι έχει τη δυνατότητα να το εφαρμόσει θα το κάνει. Και εκεί το άρθρο στη συμφωνία γίνεται υποχρέωση. Εμείς ε, το προσεγγίζουμε ως ε, μια καινοτόμο προσέγγιση σε σχέση με την προτιμησιακή ε, μεταχείριση που απλώ στο παρελθόν έδινε περισσότερο χρόνο στην αναπτυσσόμενη χώρα. Η ε, Συμφωνία Εμπορικής Ευκόλυνση θεωρείται αμοιβαία αποφελής, ένα σύνολο υποχρεώσεων και για τις ε, εκβιομηχανισμένες αλλά και για τι αναπτυσσόμενες χώρε. Ακολουθείται μη διαφορετική προσέγγιση. Πρόκειται για τελωνιακούς κανόνε και έτσι δεν αφορούν την επικράτεια ε, συγγνώμη, τους δασμούς. Επομένω, ε, το επίπεδο των δασμών μένει ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει λοιπόν απώλεια εσόδων. Όμως, Μία από τι πρώτε κινήσει για να αυξηθούν τα έσοδα μιας χώρα είναι να διασφαλίσει ότι συλλέγονται και εισπράττονται ε, οι τελωνικοί δασμοί υπάρχουν και νέες σύγχρονες μέθοδοι επίλυσης απλών ε, ζητημάτων, όπως το να έχουμε δύο ε, φυλάκια τελωνιακά σε διαφορετικές ώρες στην ίδια χώρα. Μπορεί να είναι πολύ προφανή, αλλά να έχουν τεράστια αντίκτυπο. Όταν ε, το άλλο τελωνιακό φυλάκιο είναι κλειστό, τα εμπορεύματα που ενδεχομένως ε, να λήξουν για παράδειγμα, να μπορούν έτσι να περάσουν από το άλλο φυλάκιο για να ε, εισέλθουν στη χώρα. Η σύνδεση τώρα με την TTIP. Ίσως να, μην είναι, να είναι ανόητη προσέγγιση, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια, ε, τέτοιες διατάξεις στην TTIP για τις ΕΠΑΖ. E Αυτές που έχουν συνηθεί ακολουθούν την ε, παλαιότερη προσέγγιση για την ειδική και πρωτοσιακή μεταχείριση. Εδώ έχουμε κάτι καινούριο, ένα νέο στοιχείο το οποίο γενικά μας ε, αρέσει και θα το εξετάσουμε και στη μελλοντική συμφωνία. Ήταν ε, πολυμερής προσέγγιση, ποτέ δεν την έχουμε βέβαια δοκιμάσει σε διμερείς ζητήματα. Ο κύριος Πλατών, παρακαλώ. Γενική Διεύθυνση Συνταρχών. Ναι. μου με λενε όντως. Ένα-δυο πράγματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω με βάση τα όσα ακούσαμε από τους ευρωβουλευτές. Ακούσαμε ότι οι εισαγωγέ σε αναπτυσσόμενε χώρε θα αυξηθούν. Υπάρχουν αρκετέ ε, μελέτε οι οποίε ε, καταδεικνύουν ότι οι αναπτυσσόμενε χώρε θα επιφυληθούν πολύ περισσότερο από την εφαρμογή της συμφωνίας από ότι οι ανεπτυγμένες χώρες δεν ε, περιμένουμε πολύ μεγάλη αύξηση εξαγωγών ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Υπήρξε επίσης κάποια παρατήρηση βάσει της οποίας θα πρέπει να εξετάσουμε ένα περιθώριο ευελιξίας ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες η βοήθεια που έχουμε προγραμματίσει να παράσχουμε με βάση τη Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίες ε, βασίζεται κυρίως στη ζήτηση. Ε, δεν επιβάλλονται αυτά τα 400 εκατομμύρια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, πρέπει να κοινοποιήσουν, όπως είπε ο συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, και εμείς από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε με τον τρόπο που το επιθυμούν. Μπορούμε να τους κατευθύνουμε με τη χρηματοδότηση, με τεχνική συνδρομή και δημιουργία δυνατοτήτων, ώστε να αντοπίσουν και τις αδυναμίες ε, του ιστορικού του συστήματος, ε, για να υπάρχει και αποτελεσματική εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Αυτά ήθελα να πω μόνο τώρα. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νόιζερ, έχετε να προσθέσετε κάτι. Σημείωσα τα σχόλια και θα τα διαβιβάσω στον συντάκτη των γνωμοδοτήσεων. ο κύριος Μία πρόταση επί της διαδικασίας ε, για αυτές τις συμφωνίες στο μέλλον. Τα 400 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ε, φαντάζομαι επιλέξιμα βάσει του τίτλου δημόσιας ε, επιχορήγησης για την ανάπτυξη. Θεωρούνται λοιπόν επιλέξιμα σε αυτό τον τίτλο του προπολογισμού. Εγώ θα ήθελα στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και πιο συγκεκριμένη η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να μας δίνει την αξιολόγησή της για τις ε, συνέπειες ε, των ε, ε, ποσών αυτών για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρότασή μου. Τώρα βέβαια αν εσείς έχετε την αξιολόγηση θα μπορούσατε να μας τη διαβεβαιάσετε, αλλά θα ήθελα να ξέρω τον τρόπο με τον οποίο έχουν κατανεμηθεί οι πόροι και πώς θα χρησιμοποιούνται. Κύριε Πλατών, φαντάζομαι ότι η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ κάνει μια αξιολόγηση του πώς δαπανούνται τα κονδύλια αυτά. Το ερώτημα είναι μπορείτε να τα πείτε εδώ στην Επιτροπή. Ε, κύριε Γκέρενς, ίσως αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε εμείς από πλευράς Επιτροπή είναι να εξετάσουμε τη γενικότερη εικόνα του εμπορίου και της πρόσβασης που υπάρχει, γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία συζητούμε, ε, γίνονται κάποιες αλλογές ε, στον τρόπο με τον οποίο έχουν πρόσβαση στα κονδύλια, ε, και καλό θα ήταν να τα συζητήσουμε συνολικά. Αντί να μιλάμε για πράγματα εμβαλωματικά, καλότερα θα ήταν να δούμε γενικότερα πώ έχουν πρόσβαση τα κονδύλια αυτά οι αναπτυσσόμενε χώρε και να τα δούμε. Θα το συζητήσουμε και στου συντονιστέ ίσω τι επόμενε εβδομάδε, να το εξετάσουμε ω θέμα συζήτηση στην Επιτροπή μα κάποια στιγμή στο μέλλον. Διότι εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων καθόλου επί του ζητήματο και θα ήταν χρήσιμο να έχουμε όλοι μια γενικότερη εικόνα θεμάτων πρόσβαση στην αγορά. Ίσως θα μπορούσε όμως να απαντήσει και η Κομισιόν ε, για το θέμα της ε, αξιολόγησης. Πράγματι, όσον αφορά στην αξιολόγηση, θέλω να πω ότι η Κομισιόν αξιολογεί τις εμπορικές διευκολύνσεις και αυτές πρέπει κανείς να τις αντιμετωπίζει ως τμήμα της ευρύτερης πολιτικής ε, βοήθειας, πολιτικής ενισχύσεων που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη την G20 στην Κορέα πριν από μερικά χρόνια δεσμεύτηκαν να προσφέρουν τουλάχιστον 8 δις κάθε χρόνο με τη μορφή βοήθειας, εμπορικής βοήθειας. Για να δούμε τώρα κατά πόσον καλύπτονται αυτές ε, οι υποσχέσεις ε, κάθε χρόνο κάνουμε μια αναθεώρηση της εμπορικής βοήθειας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Προσλαμβάνουμε συμβούλους οι οποίοι εξετάζουν ακριβώς το τι έχουμε κάνει στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής βοήθειας. Τώρα, ως Επιτροπή για τις εμπορικές διευκολύνσεις. Εκεί θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία για να καλύψουμε και αυτές τις υποχρεώσεις μας. Πάντως εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε χρόνο επανεξετάζουμε την κατάσταση για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε, σε ποιο μέρος του κόσμου, εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα. Κάθε χρόνο εκδίδεται μία έκθεση γύρω στο Μάιο-Ιούνιο. Νομίζω ότι σωστά θέλετε να θέσετε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, διότι θα έτσι θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα τι ακριβώς θέλουμε να ζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα μια ε, εκ των προτέρων αξιολόγηση. Συγγνώμη, πριν ε, ε, ψηφίσουμε, να ξέρουμε λίγο ποιοι είναι οι στόχοι, ποιος είναι ο τρόπος που το κάνουμε και από εκεί και πέρα τι συνέπειες θεωρεί η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ότι υπάρχουν στις χώρες ε, που είναι αναπτυσσόμενες και ποιε θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες ε, όταν δεν δίνεται αυτή η χρηματοδότηση στι αναπτυσσόμενε χώρες, διότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το εμπόριο χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια ε, για τη μείωση τη ένδυα. Ευχαριστώ. Θα το θέσουμε στην ίδια διάταξη, θα βρούμε έναν τρόπο για να γίνει αυτή η συζήτηση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τι δύο νομοδοτήσεις είναι αύριο μέχρι τι 2. Για την πρώτη σύσταση είναι να ψηφίσουμε ναι. Τους συνεργούς που θέλουν να πούν όχι. Και η δεύτερη είναι κανονική ε, γνωμοδότηση. Μπορεί να τροποποιηθεί ω συνήθω. Μέχρι τι 4 λοιπόν αύριο το απόγευμα. Και θα ψηφίσουμε στι 23 Ιουνίου. Τώρα συνάδελφοι α περάσουμε στο σημείο 9 συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για την Επιτροπή Αλίας, ε, την πρόταση απόφασης ε, για την συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό των ελευτικών δυνατοτήτων με τη Δημοκρατία της Γουινάς Μπισάου. Η προηγούμενη κοινή αλληλευτική πολιτική είχε αποφασιστεί στο τέλος της προηγούμενης θητείας και έτσι αυτές οι συμφωνίες πρόσβαση στις αλληλευτικές δυνατότητες είναι πολύ πιο φιλικές προς την ανάπτυξη και έχουν και τέτοιε αναπτυξιακές πτυχές. Γι' αυτό αποφασίσαμε να εκδώσουμε ε, γνωμοδότηση, να εκπονήσουμε γνωμοδότηση για κάθε μία από αυτές τις συμφωνίε. ούτω ώστε ε, να εκπληρούνται και ο στόχος τη μεταρρύθμισης της κοινής ελευθερικής πολιτικής. Και εγώ είχα εξηγήσει ε, στους συναδέλφους ότι πραγματικά συνεργαζόμαστε ε, στενά επ' αυτού. Ο κύριο Ντέβα είναι εισηγητή, δεν παρίσταται σήμερα και μου είπαν ότι θα τον αντικαταστήσει ο κύριο Λούκα από την ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, αλλά ούτε ο κύριο Λούκα είναι εδώ, δεν τον έχουμε βρει ακόμα ή μάλλον είναι σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο σε εισηγητή, θα δώσουμε το λόγο όμως σε σκιώδης. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος ε, θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Ο κύριος Πάγκα. Α, μόλις φτάσατε την καλύτερη στιγμή. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παρέμβω, παρότι ο συνάδελφος Δέβα δεν είναι εδώ, ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους ε, του ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντέβα για όλα όσα έχει κάνει. Σημερίζομαι τα συμπεράσματά του και θεωρώ ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτό το νέο πρωτόκολλο που προσφέρει πραγματικές ε, νέες δυνατότητες ανάπτυξης στη Γουινάμπισάου. Θα καταθέσω τροπολογίες για να υπενθυμίσω ε, δύο ζητήματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτον είναι η ανάγκη συστηματικών εκθέσεων σε ό,τι αφορά τον ε, κλάδο και τη στήριξη του κλάδου της αλίας αναφέρεται ένα σημαντικό ποσό, 3 εκατομμύρια το χρόνο και πρέπει να έχουμε ε, περαιτέρω πληροφορίες για την αξιοποίηση των πόρων αυτών. Δεύτερον, πρέπει να επιμείνουμε στην χρηστή διακυβέρνηση και την ε, καταπολέμηση της διαφθοράς ε, στην Γουινέα Μπισάου. Η ανάκληση της υφιστάμενης συμφωνίας κατόπιν του πραξικοπήματος του 2012 μας επιβάλλει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πόγκα. Τώρα είδα ότι ο κύριος Λούκα ήλθε από την άλλη επιτροπή, είναι μαζί μας. Μέχρι να καθίσει λοιπόν, σας ευχαριστούμε γιατί ξέρω ότι και εμείς ε, κινούμαστε αρκετά γρήγορα σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος συνάδελφος που να θέλει να πάρει τον λόγο. Είστε έτοιμος κύριε Λούκα είπαμε ότι ο κύριος Ντέβα σα ζήτησε να τον εκπροσωπήσετε. Σα ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε εδώ σήμερα και μετά θα δώσουμε το λόγο στου άλλου συναδέλφου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όπως είπατε ήδη, εδώ μιλώ εξ ονόματος ε, του Νέιτ Ντίβα που δυστυχώς ε, δεν κατάφερε να παρευρεθεί. Τον αντικαθιστώ λοιπόν και μπορώ να πω ότι και εκείνο αλλά και εμεί ω πολιτική ομάδα είμαστε ικανοποιημένοι από τι θετικέ πολιτικέ εξελίξει στη Γουινέα Μπισάου μετά τι προεδρικέ εκλογέ το 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακτήσει την εταιρική σχέση και τη συνεργασία μάλλον με την Γουινέα Μπισάου και επανεκκίνησε τι διαπραγματεύσει ό,τι αφορά την Συμφωνία λευτικών Δυνατοτήτων. Προβλέπονται λοιπόν ελευτικές δυνατότητες για τα ευρωπαϊκά σκάφη σε αποκλειστικές ζώνες της Γουνιάς Μπισάου για τον ε, τόνο, ε, τις γαρίδες και τα κεφαλόποδα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία, αυτό το πρωτόκολλο μάλλον για τη Γουνιά Μπισάου και από οικονομική σκοπιά. γιατί ε, φτάνουμε στα 9 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για μια τριετή περίοδο και βεβαίω ότι αφορά την ανοικοδόμηση ε, του αλευτικού κλάδου, ανάπτυξη της τοπικής αλληλεία αλλά ωφέλη προς ε, τους αλληλείς και εξαγωγές αλληλευτικών προϊόντων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι υποφελής η συμφωνία. Θα θέλαμε στο ε, σχέδιο γνωμοδότηση να υπάρξει συνένεση προς την σύνευση αυτού του πρωτοκόλου και να τονίσουμε δύο ακόμα ζητήματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γουινέα θα πρέπει να ε, βελτιώσουν τη συνεργασία και να καταπολεμήσουν την λαθρέα αλία ε, με την χρήση ειδικών ε, συστημάτων παρακολούθησης ε, δορυφορικών και το καθεξής και δεύτερον είναι σημαντικό για την εφαρμογή της συμφωνίας να αυξηθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση πόρων για την κλαδική αλία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της τοπικής αλίας και των κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Κατά τα άλλα, και μεταποίησης μάλλον. Ευχαριστούμε και στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χόιμπουκ έχει το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δυστυχώς δεν ακούμε. Δεν έχει το μικρόφωνο ανοιχτό η ομιλήτρια. Το μικρόφωνο της αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήστε λοιπόν από την αρχή. Εμείς οι πράσινοι δεν θα εγκρίνουμε την συμφωνία και θα σε εξηγήσω γιατί. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκε χωρίς να υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις και όπως αναφέρθηκε με βάση το κείμενο του 2012. Οι διαπραγματεύσεις για το πρωτόκολλο διεκόπησαν το 2012 με το πραξικόπημα και μετά ξανάρχισαν ακριβώς εκεί που είχαν σταματήσει. Και μάλιστα Κατά την άποψή μου ε, χρησιμοποιήθηκε το απαρχιωμένο πλέον κείμενο, δηλαδή ε, τα λιεύματα και όλα τα παλιά στοιχεία χωρίς να γίνει καμία νέα αξιολόγηση. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, το πρωτόκολλο αυτό δεν συμβατίζει με την ε, κοινή ελευτική πολιτική, κάτι το οποίο, μια πολιτική η οποία τέθησε ισχύ το 2014. Επίσης ε, γίνεται λόγος για πλεονάζουσες ε, αλλιευτικές μεθόδους και πλεονάζοντες πόρους. Αυτοί όμως πρέπει καταρχήν να διαπιστωθούν. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα με, το, με τα αλλιεύματα. Όχι να δουλεύουμε με τα στοιχεία του 12. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση θα χρειαζόμασταν μια επιστημονική μελέτη για να μας ε, δει τι ακριβώς γίνεται με τα αλλιεύματα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν με άλλες μεταναστευτικές κινήσεις των ψαριών και για όλα αυτά εμείς δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Επίσης δεν υπάρχει διαφάνεια για την πρόσβαση από άλλους αλλοδαπούς στόλους. Ε, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η αλία γίνεται μόνο από ευρωπαϊκούς στόλους, γίνεται και από ασιατικούς και από ρώσικους, γιατί υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γουινέα Μπισάου. Και εκεί λοιπόν δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι δικές τους οι ποσοστώσεις, ποιες είναι οι ποσοστώσεις της, Κίνα, της Κίνας που το 2014 εκείνη ήταν παρούσα με δύο σκάφη. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα στοιχείο για τα λιεύματα και επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτό δεν συμβαδίζει με τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό που είπε ο κ. Λούκα, δηλαδή η τομεακή βοήθεια ήτια 2,9 ε, εκατομμύριο το χρόνο πρόκειται να εκταμιεύονται όμως ε, το Υπουργείο μόνο του δεν έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει αυτά τα κονδύλια. Εντάξει να τα πάρουν μπορούν είμαι σίγουρη αλλά το τι θα τα κάνουν περί αυτού πρόκειται. Το Υπουργείο λοιπόν δεν έχει την απαραίτητη υποδομή και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να εκταμιευθούν κονδύλια και σε άλλα Υπουργεία ή σε ΜΚΟ. Δεν έχει όμως ληφθεί απόφαση και γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει σαφήνεια πριν προχωρήσουμε στην υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ο κύριος Τζέλα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πριν συμφωνήσω σε μια τέτοια συμφωνία, έχω και εγώ περίπου τις ίδιες ερωτήσεις όπως και η κυρία Χόιμπουχ. Η πολιτική κατάσταση στη Γουνέα Μπισάου, ναι μεν, μετά τις εκλογές, από το 2014 και μετά, και εφ' εξής δηλαδή, ε, η κατάσταση είναι πιο δημοκρατική, εντάξει μέχρι τότε υπήρχε δικτατορία, Ας το δεχτούμε αυτό, Ξεκολουθεί όμως να υπάρχει αστάθεια και αυτό που ενδιαφέρει εδώ κυρίως είναι τα παράκτια ύδατα μπροστά από την Γουνεαμπισάου, κυρίως γενικότερα τα παράκτια ύδατα στη Δυτική Αφρική. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι εκεί υπάρχουν ε, μεγάλες ποσότητες ψαριών από τη Δυτική Αφρική μέχρι τις Κανάριες νήσους. Εν τω μεταξύ όμως ε, πάρα πολλά είδη ψαριών βρίσκονται υπό απειλή, κινδυνεύουν. Εν τω μεταξύ πάρα πολλά κράτη αλλιεύουν τόπου, εξαντλούν τις ε, τοπικές θάλασσες και οι ντόπιοι τίποτα πια να ψερέψουν. Αποτέλεσμα αυτού είτε γίνονται πειρατές ή έρχονται στην Ευρώπη ως πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κάνω μία ερώτηση. Η Κομισιόν λέει ότι αν υπογράψουμε μία συμφωνία εμείς θα ψαρεύουμε μόνο το πλεόνασμα των ψαριών με τα σκάφη μας. Αυτό τώρα το πλεόνασμα πώς μπορεί κανείς να το διαπιστώσει. Πώς θα μπορεί να πει με σιγουριά ότι αυτό είναι το πλεόνασμα που περισσεύει και στο ψαρεύουν οι Ευρωπαίοι. Κανείς, ε, κάνοντας αυτήν την ερώτηση, κανείς δεν μπόρεσε να μου δώσει μια λογική απάντηση. Και από την άλλη βλέπουμε περίπου 500 κινέζικα σκάφη ε, να βρίσκονται επιτόπου και από την Ταϊβάν και από την Ιαπωνία και από άλλα κράτη. Σοβιετικά, Ουκρανικά, Λιθουανικά, Λετωνικά, όλα αυτά σκάφη βρίσκονται επιτόπου Βέβαια όχι με δική τους σημαία, αλλά με σημαίες δυτικοαφρικανικών κρατών, τις οποίες τις ε, προμηθεύτηκαν και ψαρεύουν αυτοί ως να ήταν ε, γηγενείς, που δεν είναι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε κατά την άποψή μου μία σε βάθος αξιολόγηση του τι ακριβώς διαδραματίζεται στις ε, ακτές της Δυτικής Αφρικής. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις ε, ποσότητες και για τα λιεύματα επιτόπου και το επόμενο που χρειαζόμαστε ε, για το υποτιθέμενο πλώνισμα μίλησα. Ε, το άλλο που θέλω να πω είναι ποιος είναι ο δικαιούχος από όλους εμάς και πώς ελέγχεται. Ποιος είναι εκείνος ο, ο οποίος ψαρεύει επί τόπου, με τι προδιαγραφές, πού εκφορτώνει τα ψάρια του, γιατί ο τόνος, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι επιθυμητός μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού και πουλιέται μάλιστα με τιμές ρεκόρ. Ελπίζω λοιπόν να μην καταλήγει τελικά ε, ακριβώς εκεί που είναι ιδιαίτερα επιθυμητός και χωρίς ε, ελέγχους ενώ από την άλλη πολλοί προσπαθούν να εφαρμόζουν βιώσιμες αλληλευτικές μεθόδους. Αυτά είναι ερωτήματα ε, που θα ήθελα να ξεκαθαριστούν πριν τελικά συμφωνήσουμε για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Και κατά τα άλλα, εντάξει, κατανοώ, ε, είναι, μεγάλα, είναι πολλά τα λεφτά για μια μικρή χώρα ε, και τα χρήματα τελικά πράγματι πρέπει να βοηθήσουν τους ντόπιου. Σε ποιον λοιπόν θα χορηγήσουμε τα χρήματα μπορεί να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος έτσι ώστε τα υποεκταμείευση κονδύλια τελικά να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που εκταμιεύονται, δηλαδή για να τονώσουν την τοπική οικονομία και κυρίως ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι ερωτήματα που έχω, δεν βρίσκω τις απαντήσεις ε, στη συμφωνία και γι' αυτό λοιπόν ε, έχω θέσει αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ, εσείς έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση για το θέμα της ε, τομεακής βοήθειας του προπολογισμού. Ποιοι ήταν οι όροι της συμφωνίας που οδήγησαν ε, στη βοήθεια αυτή προς την ε, Γουινέα. Ε, πώς ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γιατί τους δίνεται αυτή η τομεακή βοήθεια και επίσης όσον αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία, είναι θέμα στρατηγικής σημασίας. Ποιος την οργανώνει αυτή την εποπτεία. Κατά την άποψή μου αυτή θα πρέπει να γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι εκχωρείται στα ε, κράτη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια σύμπραξη. δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν από 10 χρόνια δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που ήταν αρμόδια. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κάποιος άλλο το λόγο. Θα... θα δώσω το λόγο στον κύριο Εμμάνουελ Μπέρκλey από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ Ίσως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε και κάτι στην Επιτροπή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό το συγκεκριμένο ποσό προς την ε, κυβέρνηση της Βουινέα Μπισάο. Τι ε, συνεισφορά ε, ε, ε, έχει ο ιδιωτικός τομέας, αυτοί που αλλιεύουν και εκμεταλλεύονται τα αλλιεύματα. Ε, υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο επιστρέφεται στους φορολογουμένους. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, ε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να μεταρρυθμίσει την κοινή ελευθερική πολιτική περισσότερο από ό,τι συμφωνήθηκε τελικώς. Και εμείς ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν συμφωνήσαμε και εμείς θεωρήσαμε περισσότερο. Το θέμα είναι ποιο πληρώνει. Πληρώνει ο φορολογούμενος, αλλά τα ωφέλη οι επιχειρήσεις αν δεν κάνω λάθος δεν πληρώνουν τίποτα. Δεν είμαι βέβαιη ότι πληρώνουν κάτι για να λάβουν τις άδειες. Ε, ξέρω ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή και ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση Μάρε ε, γνωρίζει αυτά τα ζητήματα. Ε, εσείς είστε ορμόδιος για τη Γενική Διεύθυνση Μέρη. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους ε, κυρίους και κυρίες ευρωβουλευτές που εξέφρασαν την άποψή τους για το πρωτόκολλο αυτό. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρωτόκολλο για μας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά από ε, οικονομική σκοπιά, ε, διότι συνεισφέρουμε με 9 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια αλλιευτική συμφωνία που αφορά και μια σειρά από αλλιεύματα και διάφορα είδη, Επομένω, είναι αρκετά μεγάλο ενδιαφέροντο για το στόλο μας και είναι μια μεικτή συμφωνία όπως την αποκαλούμε, μια αντίστοιχη με αυτή που έγινε με το ε, Μαρόκο, και ε, υπάρχουν αρκετά ωφέλη για αρκετούς οικονομικούς φορείς. Ε, βέβαια αυτό το ποσό είναι και σημαντική συνέπεια για τον προπολογισμό της Γουινέας Μπισάου γιατί όπως γνωρίζετε είναι μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Επομένως το ποσό αυτό το οποίο τους δίνουμε συνεισφέρει για να ξεκινήσει η λειτουργία του προπολογισμού της χώρας ε, είναι περίπου στα 9,2 εκατομμύρια και υπάρχει και καλή διαχείριση της αλληλείας με ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο καθορίζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται με τη χώρα. Θα ήθελα να προσπαθήσω τώρα να σας πω ε, κάποια στοιχεία λίγο πιο αναλυτικά όσον αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν. Καταρχάς, ε, όντως πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι το 2012 έγινε διαπραγμάτευση με τη Βουινέα Μπισάου, είμαστε στο 2015, ε, έχουν περάσει λίγα χρόνια, υπήρξε μια διακοπή που οφείλονταν στην ε, πολιτική κρίση που έπληξε τη χώρα. Γιατί δεν έγινε νέα διαπραγμάτευση. Ε, είχαμε φτάσει στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις μας είχαν οδηγήσει σε μονογραφή ενός κειμένου και αν έπρεπε να ξαναγίνουν να διαπραγματεύσει θα έπρεπε να ξεκινήσουν όλα από την αρχή, να γίνει μια νέα αξιολόγηση, μια νέα εντολή του Συμβουλίου και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης αρκετών μηνών. Θα είχαμε χάσει λοιπόν πολύτιμο χρόνο για το στόλο μας, ο οποίος ήταν αναμονή των αδειών για να ξεκινήσει αλία, αλλά και απώλεια και για τη Γουινέα Μπισάου, ε, που θα έχανε κάποιου σημαντικού οικονομικούς πόρους. Βέβαια, η ανησυχία για την κατάσταση των αποθεμάτων είναι μια συνεχής ανησυχία και πάντα τη λαμβάνουμε υπόψη μας όταν συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες ελίας. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις το 2012 χρησιμοποίησαμε τις καλύτερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υπενθυμίζω ότι είναι γνωμοδοτήσεις οι οποίες διατίθενται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλίας όπως για παράδειγμα τη ΕΚΑΦ που είναι υπό την αιγίδα του ΦΑΟ ε, αφορά τη συγκεκριμένη χώρα αλλά και άλλες χώρες λοιπόν η συγκεκριμένη περιφερειακή εργόνωση. Ε, είχαμε λάβει υπόψη μας λοιπόν τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και είχαμε και κάποιες προσωπικές ανησυχίες γιατί είχαμε αποφασίσει να μειώσουμε τον αριθμό των επιτρεπόμενων αλευμάτων. Ε, λάβαμε υπόψη μας και κάποια τεχνικά μέτρα όπως για παράδειγμα το μέγεθος των ματιών του δικτύου. και υπάρχει ένα διάστημα το οποίο δεν θα θέλαμε να χαθεί ε, γιατί θα έπρεπε να περιμένουμε για να λάβουμε καινούργιε ε, επιστημονικέ γνωμοδοτήσει. Είναι ένα τρόπο να βοηθήσουμε τη Γουινέα Μπισάου, να του δώσουμε κάποια πυρογνωμοσύνη και να μπορέσουν να κάνουν κάποιε συμφωνίε αλληλεία και να λάβουν και αυτή τη σημαντική χρηματική βοήθεια για την εποπτεία. Αντί λοιπόν να είμαστε απόντε και να αφήσουμε τα ε, δυνατότητα σε άλλου στόλου, παραδείγματο χάρη ασιατικού στόλου, προτιμήσαμε να είμαστε εκεί ω παρόντε και να βοηθήσουμε για την εκμετάλλευση των πόρων του. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να ενισχύσουμε στο νέο πρωτόκολλο τις δυνατότητες της κοινή μεικτής ε, επιστημονικής επιτροπής ε, που ε, συστήθηκε με τη χώρα αυτή και αυτό το οποίο κάναμε από τους πρώτους μήνες ισχύω του πρωτοκόλλου είναι να συναντηθεί αυτή η μεικτή Επιτροπή που περιλαμβάνει επιστήμονες και από τη Γουινέα Μπισάου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Απρίλιο και τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι ότι υπήρχε μια σταθερή αλλιευτική προσπάθεια από το 2010. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή για τα είδη τα οποία αλλιεύονται στη Γουινέα Μπισάου. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία και για την αλλιευτική προσπάθεια και για την παρουσία ασιατικών στο, ε, στόλων ε, Έχουμε μια σαφή εικόνα για τον αριθμό των σκαφών που αλλιεύουν, ε, τι κατηγορία είναι, τι ήδη αλλιεύουν και αυτό φυσικά ε, μας οδηγεί και σε συμπεράσματα για το τι συνέπειες υπάρχουν για τα αποθέματα. Και σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον επιστημονικό διάλογο με τη Γουινέα Μπισάου, ε, βοηθώντας τους ταυτόχρονα για να εφαρμόσουν μέτρα και σε στατιστικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης και εποπτείας, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Έχουμε επίσης, όπως σας έλεγα, ένα πρόγραμμα δράσης, ε, τη λεγόμενη τομεακή στήριξη. Πρόκειται για μια στήριξη στον προϋπολογισμό, η οποία περιλαμβάνει και μια σειρά από δράσεις, οι οποίες στόχο έχουν να βελτιώσουν τη ε, διαχείριση της αλίας. Παραδείγματος χάρη ε, χρηματοδότηση κάποιων υποδομών, ε, ε, αυτό έγινε με βάση το προηγούμενο πρωτόκολλο, αλλά υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχουν κάποιες υποδομές, υπάρχουν κάποιες αναλύσεις σε υγειονομικό επίπεδο, ε, γίνονται σε εργαστήρια. Στο προηγούμενο πρωτόκολλο είχαμε χρηματοδοτήσει τα εργαστήρια, τώρα χρηματοδοτούμε τον εξοπλισμό των εργαστήριων. Πρόκειται λοιπόν για μια στρατηγική, η οποία είναι αρκετά συνεπής από πλευράς Γουινέα Μπισάου, για να μπορέσει να ε, αξιολογήσει τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους και να μην δίνει απλώς άδεια σε κάποια σκάφη να έρχονται να λεύουν και να φεύγουν, αλλά να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές ε, και για μεταποίηση ελευμάτων που είναι ε, και τομέας ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και φυσικά και δυνατότητες εξαγωγών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο θέμα επί του οποίου επιμείναμε στο πρόγραμμα δράσης το οποίο καθορίστηκε με τη Γουινέα Μπισάου είναι η εποπτεία των υδάτων τους φυσικά ε, διότι υπάρχουν αρκετοί ε, παράγοντες, αρκετές δυνάμεις αν θέλετε που είναι παρούσες και ε, υπάρχει το εξής, ε, ε, η λειτουργικότητα του συστήματος VMS, του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης των σκαφών. Αυτό το χρηματοδοτήσαμε, θα συνεχίσει η χρηματοδότηση ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό και λογικά μέχρι το τέλος του 2015 θα έχει τους πρώτους, τα πρώτα αποτελέσματα αυτό το σύστημα και θα μπορεί η Γουινέα Μπισάου να παρακολουθεί και τα λευτικά σκάφη της χώρας της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στα ύδατα αυτά. Θα μείνουμε στον τομέα αυτό, το είπατε κι εσείς, υπάρχουν αρκετά χρήματα. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν θέματα απορρόφησης, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε επίσης να ενισχύσουμε και τα, ε, τα, τις διάφορες προσπάθειες επιτήρησης Όσον αφορά την εραστική αλληλεία, να σας πω και δύο λόγια, γιατί και αυτό είναι συστατικό στοιχείο της, ε, του προγράμματος δράσης μας. Υπάρχουν μια σειρά από δράσεις για να χρηματοδοτήσουν, να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό των αλλιέων ε, από τη Γουινέα Μπισάου. Επίσης ε, αγορά εξοπλισμού ασφαλείας, να γίνει καταγραφή των διαφόρων σκαφών, πυρόγες και ό,τι άλλο υπάρχει και να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν και να μπορέσουμε να έχουμε και ε, μια δραστηριότητα για αυτούς τους αλείς που ζουν από τη θάλασσα στη Γουινέα Μπισάου. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, έχουμε τακτικά αυτές τις μικτές επιτροπές που είναι ε, ένας, ε, ένα βήμα διαλόγου με τις χώρες αυτές. Μία φορά το χρόνο σίγουρα, σε κάποιες περιπτώσεις σε μικτές συμφωνίες συναντιούνται και περισσότερες φορές, όπως συμβαίνει και με τη Γουινέα Μπισάου. Τον Ιανουάριο ε, εγκρίναμε ένα πρόγραμμα δράσης στην πιο πρόσφατη συμφωνία, ε, υπευλήθηκε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η προσπάθεια που κάνουμε για να δούμε με τις υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες και με τη βοήθεια της Αντιπροσωσμίας Επιτόπου και της ε, Αλλιευτικής Επιτροπής που, που εδρεύει στον Ντακάρ, να δούμε εάν εφαρμόζονται όλα τα στοιχεία. Ε, επαγρυπνούμε για να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν αποτέλεσμα, αν υπάρχουν συγκεκριμένε συνέπειε. Ε, ελπίζουμε ότι θα υπάρχει επιτυχία και θα υπάρχουν ε, αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε αυτό που είχαμε προβλέψει. Το 2011 υπήρχε ένα πρωτοκόλλο επίσης ε, ε, ενισχύ με τη Γουινέα Μπισάο. Δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτά που είχαν γίνει τότε και αποφασίσαμε να μειώσουμε εκ των προτέρων την χρηματοοικονομική συνδρομή που δίναμε στην τομέα και ανάπτυξη. Έχουμε δηλαδή μέσα πίεσης, έχουμε μέσα τιμωρητικά και επαγρυπνούμε και μπορεί να είναι λίγο ε, παροχημένο το πρωτόκολλο, αλλά και τότε είχαμε συμπεριλάβει και αρκετά θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση των αλλιευτικών συμφωνιών για παράδειγμα τη ρήτρα αιρεσιμότητας, η οποία επιτρέπει να μειώσουμε ή να αναστείλουμε τις ε, χρηματοδοτήσεις της ε, τομεακής στήριξης. Επίσης, η συμφωνία αυτή, παρά το γεγονός ότι μονογράφηκε το 2012, είναι αρκετά σύγχρονη. Υπάρχει ρήτρα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ρήτρα διαφάνειας, ρήτρα μη διάκρισης μεταξύ των στόλων μας ή άλλων στόλων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε αυτό το νέο πρωτόκολλο να τεθεί σε ισχύ διότι υπάρχει εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές, πρέπει να τις βοηθήσουμε και να παρακολουθούμε η διεισόμαση τι ακριβώς γίνεται στη Γουινέα Μπισά. Νομίζω ότι απάντησα σε αρκετέ ερωτήσεις και επίση υπήρχε και μια σαφέστατη ερώτηση για το πώς ε, έγινε η παρακολούθηση ε, των χρημάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση. Υπάρχει το ένα τμήμα που αφορά την τομεακή στήριξη, λοιπόν, τη θέμα της διαχείρισης της αλληλείας, που είναι αυτά τα οποία σας ανέπτυξα λίγο πιο διεξαδικά. Και μετά υπάρχει το μεγαλύτερο τμήμα, 6, 6 εκατομμύρια ευρώ συγγνώμη, το χρόνο, ε, τα οποία είναι και λίγο το πνεύμα των συμφωνιών μας, είναι εμπορικές συμφωνίες, ε, και ίσω δεν ζητούμε και τόσε λεπτομέρειε και εξηγήσει για το τι ακριβώ γίνεται με αυτά τα χρήματα. Πηγαίνουν στον προπολογισμό του κράτου. Ε, ξέρω βέβαια ότι υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης και πλαισίασης της Γουινέα Μπισάου που γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ μαζί με την στήριξη στον προπολογισμό και γίνεται και από τους ε, ε, συναδέλφους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, επομένως το ποσό αυτό πηγαίνει στο κρατικό κορβανά ε, και από εκεί και πέρα ε, τα θεσμικά όργανα ε, παρακολουθούν τη χώρα για να μπορεί να ξεφύγει από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει και αυτοί παρακολουθούν και το τι γίνεται με τα χρήματα αυτά που μπαίνουν στον προπολογισμό τους. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε και για να απαντήσουμε και στην ερώτηση της Προέδρου ότι υπάρχει συνεισφορά των πλειοκτητών στις τελευταίες διαπραγματεύσεις αυξήσαμε κατά 25% την ε, συνεισφορά που πληρώνουν οι πλειοκτήτες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αλληλευτική συμφωνία. Δεν μπορώ να σας δώσω ένα ακριβές ποσό, διότι το ποσό το οποίο καταβάλλεται εξαρτάται από τον αριθμό των αδειών, από τη δραστηριότητα, από τα αλλιεύματα. Είμαστε στο πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλου. Ε, μάλλον προς το τέλος του έτους, ε, στην επόμενη μεικτή επιτροπή θα μπορούμε να κάνουμε έναν απολυγοσμό των οικονομικών εσόδων που είχαμε από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει όμως συνεισφορά τους και η συνεισφορά των πλειοκτητών ε, θα θέλαμε να είναι το μεγαλύτερο τμήμα ε, σε σχέση με τον προϋπολογισμό το δημόσιο που δίνεται και επιβαρύνει τους φορολογουμένους. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Να πω και κάτι επιπλέον. Πέραν της συμφωνίας υπάρχει και τεχνική συνδρομή ε, προς τη χώρα. Οι υπηρεσίε τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΑ και ο Οργανισμό Ελέγχου τη Ελίας, το ΒΙΚΟ και η Διεθνή Ομάδα του παρακολουθεί. Υπάρχουν επίση ε, σχέδια για μία αποστολή στου επόμενου μήνες στη Γουινέα Μπισεωά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι σε επίπεδο ελέγχου αλληλεία χρησιμοποιούνται καταλήλω αυτά τα κονδύλια, ότι λειτουργεί το σύστημα VMS για την παρακολουθήση των σκαφών, ότι το σύστημα ώρες ε, ε, για την αυτόματη δήλωση των αλλιευμάτων θα εγκατασταθεί και αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από δράσεις που προβλέπονται από αυτό το πρωτόκολλο. Πρόκειται για ένα σημαντικό εταίρο, ευάλωτο μεν, αλλά πολύ σημαντικό και με πόρους που αξίζουν τον κόπο να δημιουργήσουμε κατάλληλες δυνατότητες, να αναπτύξουν οι ίδιοι τις δυνατότητές τους που θα ξεκινήσουν μετά από κάποιους μήνες και θα ε, ισχύουν για όλη τη διάρκεια ζωής του πρωτοκόλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λούκα, θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι ουσιαστικά. Δυστυχώ δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε ερωτήματα. Όμως σημειώνουμε τα όσα έχουν υποθεί και θα τα διαβιβάσουμε στον εισηγητή και εκείνος θα απαντήσει προσωπικά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο τμήμα απλώ δίνεται συνένεση της νομοδότησης ή την απορρίπτουμε. Και δεύτερον έχουμε ε, πρόταση ψηφίσματος. Στο πρώτο τμήμα μπορείτε μόνο να πείτε το αντίθετο από αυτό που λέει ο συγητής. Και η προθεσμία κατά των απολογίων είναι αύριο μέχρι τις 5 το απόγευμα και για τα δύο τμήματα της πρότασης. Για το πρωτόκολλο με την Γουινέα Θα ψηφίσουμε σε μερικά λεπτά. Όμω, επειδή είπαμε 5 και 4, θα ήθελα να επιστρέψω στι ε, ανακοινώσει. Πολλοί συνάδελφοι δεν ήταν εδώ στις, ε, στην αρχή τη συνεδρίαση. Να σα υπενθυμίσω, λοιπόν, για αυτήν την εβδομάδα. Ξέρετε ότι έχουμε τι ημέρε Ευρωπαϊκή Ε, Πολλά συμβαίνουν στο Τούγε Ταξί εδώ στου Βρυξέλλες. Ε, εστάλει ένα ενημερωτικό mail για να λάβετε τα διαπιστευτήρια, γιατί τα χρειάζεστε. Επομένω, αρχικά πρέπει να λάβετε αυτό το έγγραφο για να μπείτε και εμεί βεβαίω έχουμε και την ε, Πέμπτη το πρωί τη δική μα εκδήλωση. Όλοι οι ευρωβουλευτέ όμω είναι ευπρόσδεκτοι σε όλε αυτέ τι εκδηλώσει. Εάν δεν έχετε λοιπόν το πρόγραμμα και θέλετε να πάτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κριστιαν και τον Γιάσπερ. Και στους δύο λοιπόν. Ιδίω για την Πέμπτη το πρωί στις 10 παρατέταρτο. Την Τετάρτη στις 2.30 ε, έχουμε κοινή ανοιχτή ε, συνεδρίαση ε, της Επιτροπής μας με τον Γιώργο Κουτέσα που είναι πρόεδρος της Ολομέλειας του ΟΗΕ και θα έρθει γιατί ακριβώς είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτά τα ζητήματα, στα SDGs και γι' αυτό θα έρθει να μας μιλήσει. 2.30 το μεσημέρι της Τετάρτης. Και στις 6 την Τετάρτη και πάλι στο Παρλαμεντάριουμ αυτή τη φορά θα έχουμε ε, την, ε, μία έκθεση για τα οικογενειακά γεύματα. Το είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από μερικού μήνε. Αυτή τη φορά θα είναι στο Παρλαμεντάριουμ και έτσι περισσότεροι θα έχουν πρόσβαση. Έχουμε τα εγγένεια λοιπόν αυτής της έκθεσης και την 5η στις 9 το πρωί, 4 Ιουνίου, θα έχουμε μία έκτακτη ε, κοινή συνάντηση DEVA FED ε, για την ε, ανθρωπιστική αντίδραση στην κρίση στο Ιράκ. Η κυρία Καν για τα ανθρωπιστικά ζητήματα και εκπρόσωπος ε, του Ιρακινού Κοινοβουλίου, αν δεν κάνω λάθος. πρόεδρος, συγγνώμη, του Ιρακινού Κοινοβουλίου. Αυτά για την ε, Πέμπτη το πρωί και την Παρασκευή, τη Δευτέρα μάλλον, στο Στρασβούργο, 8 παρα το βράδυ, θα έχουμε κοινή συνεδρίαση ΔΕΒΕ και ελέγχου του προπολογισμού για την ε, αξιολόγηση της ε, στήριξης ΔΕΦΚΟ. Γιατί έχουν ακουστεί πολλές κριτικές και το ελεγκτικό συνέδριο έχει εκπονήσει δική έκθεση. Το πρωί λοιπόν 8 παρατέταρτο, τη Δευτέρα μάλλον, 8 παρατέταρτο, όλοι οι συνάδελφοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν σε αυτή την κοινή ε, συνεδρίαση για να εξετάσουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και θα αξιολογήσουμε ακριβώς αυτή την εκταμίευση δημοσίου χρήματο. Καλό θα ήταν να τα έχουμε όλα αυτά σε ένα σημείωμα, λοιπόν, να ζητήσω από τη συνάδελφο να το κάνει. Πού και πότε γίνεται το καθένα. Γιατί είναι πολλές αυτές ε, και οι έκτακτες ε, συνεδριάσεις και οι λοιπές εκδηλώσεις. Όλα αυτά μαζί. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανακοινώσεις. Συγγνώμη, παρατηρήσεις για τις ανακοινώσεις. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 10. εντολή για το τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό 2016. Κύριε Λίτς, θέλετε να πείτε κάτι? Αιτιολόγηση ψήφου. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Προπολογισμός 2016. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές με τους οποίους ε, συνεργαστήκαμε. Ήρθαμε σε επαφή για να βρούμε κοινό τόπο για ένα κείμενο που έχουμε, στο οποίο έχουμε καταλήξει τώρα και θα ψηφίσουμε και τις ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία. Sorry, I've just been given something to announce here. Α, τώρα μόλις μου έδωσαν κάτι το οποίο θα πρέπει να ανακοινώσω και δεν το είχα συνειδητοποιήσει αρχικά. Πιο μετά, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα το ανακοινώσω. Ωραία, θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Εντολή για το τριμερή διάλογο για το προπολογισμό 2016. Να ελέγξουμε πρώτα. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίστε ό,τι θέλετε, δεν έχει σημασία. Απλώ να ελέγξουμε ότι λειτουργούν τα μηχανήματα. 17 ψηφίσαντες. Όχι, είναι ένας απλός έλεγχος. Check everything is working. Vote is closed. Πέρας. Okay, it's working. Εντάξει, όλα καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αν ναι, πράγματι αρχίσαμε τη ψηφοφορία ένα λεπτό νωρίτερα από το προβλεπόμενο, εντάξει, πέρας ψηφοφορίας... Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Καταπίπτει. Γιατί εκείνη η τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφορία για τροπολογία 10. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τη 13 θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία. Α, είναι στο τέλος της, ε, του εκλογικού καταλόγου. Υπέρ. κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται ψηφίζουμε αρχικά την προφορική τροπολογία να ελέγξουμε έναρξη πέρας Εγκρίνεται. Έτσι κι αλλιώς. Καταπίπτει λοιπόν η 13. Γνώριζαν όλοι οι σκιώδει αυτή την προφορική τροπολογία. Έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, νομίζω. Α, εγκρίνεται. 15. Ε. Υπέρ. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε τη 17. Νομίζω εγκρίνεται. Πέρας.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 Μετά μια πολύ απλή ψηφοφορία για την ε, αλληλευτική συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη. Δεν υπάρχουν τροπολογίε ε, προ την πρόταση. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το σχέδιο νομοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη. Πέρα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια στον κύριο Μισελ παρότι δεν βρίσκεται εδώ. Τώρα περνάμε στα λίγο πιο δύσκολα. Έχω πολλές ανακοινώσεις και μετά να δώσουμε το λόγο στην Έλλη Σουλάν για να σας πει δύο λόγια. Λοιπόν, να πω τα τεχνικά πρώτα και μετά θα σας δώσω το λόγο. Λοιπόν, πρώτον, το ECR ζήτησε χωριστή ψηφοφορία σε τρεις τροπολογίες. Ήταν η συμβαστική πρόταση αρχικός, αλλά το ECR θέλει να ψηφίσουμε ξεχωριστά τώρα. 114, 15 και 67. Είναι όλε ε, στον κατάλογό σα. θα ε, ψηφιστούν ξεχωριστά, δεν θα καταπέσουν αν περάσουν οι συμβιβασμοί, ούτως ή άλλως ε, θα έχουν, φαντάζομαι, οι πολιτικές ομάδες ενδείξεις. 114, σελίδα 7. 50 και 67. Όχι 15, 50 και 67. Θα ψηφιστούν χωριστά, δεν καταπίπτουν, δεν περιλαμβάνονται στο συμβιβασμό, επομένως δεν έχουν σχέση με το αν θα περάσει ο συμβιβασμό ή όχι. Και μετά, λείπουν κάποια στοιχεία, δεν αναφέρονται πουθενά. Οι 130 των πρασίνων δεν υπάρχει πουθενά. Θα σας δώσω χρόνο τώρα, ώστε το προσωπικό των ομάδων να πει στα μέλη τους τι πρέπει να κάνουν, αν δεν υπάρχει καθόλου στον κατάλογο. Οι 130 των πρασίνων δεν ήταν στον κατάλογο ψηφοφορίας. Σα παρακαλώ συμπεριλάβετε έτσι στην σελίδα 8 μετά από την 129. Και ε, το ξέρω ότι δημιουργεί σύγχυση, θα προσπαθήσουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Από ό,τι μου λένε είναι στη σελίδα 8. 129 την έχετε λογικά και προσθέτουμε και την 130. Λείπει μία. Λοιπόν, Με άλλα λόγια, 129 και υπάρχει και μία 130 που έχει παραληφθεί κατά λάθο, θα έπρεπε να βρίσκονται στον κατάλογο των ψηφοφοριών σα. Τώρα οι ομάδε πρέπει να βρουν πώ θα ψηφίσουν, σω θα μπορούσε να του πει το προσωπικό. Ελπίζω να γνωρίζουν και να ξέρουν τι να πούνε στι ομάδε. Είναι σαφέ αυτό να ρωτάω του συντονιστέ να σα δώσω ένα λεπτάκι μπορεί να πει το προσωπικό στους συντονιστές πώς θα ψηφίσουν η ομάδα τους ε, στην ε, τροπολογία αυτή που δεν υπάρχει στον κατάλογο. Yeah, the advising Ο εισηγητής ζητά εποχή. Σωστά για την 130. Madam Rapporteur, is that correct? Η συγγήτρια δεν ξέρω αν συμφωνείτε και ε, στην 130 προτείνεται να απόσχουμε, έτσι δεν είναι. Δεν είναι στον κατάλογό σας, συνάδελφοι, συγγνώμη, θα έπρεπε να βρίσκεται στον κατάλογο. Έχετε μία επιπλέον λοιπόν τροπολογία. Δεύτερον, και άλλη τεχνική ανακοίνωση λοιπόν. Έχουμε δύο τροπολογίες στον κατάλογο των ψηφοφοριών που είναι μη παραδεκτές. Παράγραφος από τη γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ, παράγραφοι 16 και 17 της γνωμοδότησης της ΕΚΟΝ. Δεν είναι παραδεκτές ε, γιατί αφορούν την Ευρώπη και συμφωνήσαμε με την Επιτροπή ΕΚΟΝ ότι δεν θα ψηφιστούν τα θέματα αυτά, είναι θέμα δικής τους αρμοδιότητας. Γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ 13-16 είναι μη παραδεκτές γιατί δεν έχουν καμία σχέση με αναπτυξιακή πολιτική, αφορούν ευρωπαϊκή πολιτική. Τα έχετε ήδη αυτά. Ωραία. Σαφές αυτό. Να το διευκρινίσουμε λοιπόν ότι δεν είναι παραδεκτές αυτές οι τροπολογίες. Ε, ακυρώθηκαν τα Eurostar και δεν πρόλαβα να τα πω σε προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν είχα χρόνο. Η Έλλη λοιπόν η εισηγήτρια θα σας δώσει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους και για τις κοινέ μας προσπάθειες. Νομίζω ότι ψηφίζουμε ένα καλό κείμενο σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει. Σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά υπήρχε πνεύμα συνεργασίας, το οποίο θα μας επιτρέψει να εγκρίνουμε ένα πολύ φιλόδοξο και πολύ ισχυρό κείμενο της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί άριθμες τεχνικές δυσκολίες, ε, η τροπολογία 130 διαπιστώσαμε ότι έλειπε από τον κατάλογο ψηφοφορίας. Ε, όπως σα είπα, η θέση μου ως εισηγήτρια είναι να εδώ. Και τίποτα άλλο. Καλή ψήφο. Thank you. This is an report, Ευχαριστώ. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση, συνάδελφοι, διότι ε, θα αφορά και το τμήμα των εργασιών μας όταν θα πάμε στην Αντίσα Αμπέμπα και θα έχουμε την αντιπροσωπεία μας για τα αναπτυξιακά ζητήματα. Θα έχουμε λοιπόν ε, και αυτό το, έγγραφο που θα προσθεθεί στην έκθεση για την ανάπτυξη που προσθέσαμε πριν από δύο εβδομάδες. Έχουμε λοιπόν την έκθεση για τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή της κυρία Σλάιν και ξεκινούμε με τη συμβαστική πρόταση 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 στην επόμενη σελίδα απευθείας. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88, παράγραφος 3. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 92. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24. Καταπίπτουν αρκετές υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία στην 109 της παραγράφου 6. Υπέρ. Χωριστά ψηφίζουμε την 109 παραγράφου 6 του κυρίου Λούκε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 114. Πάλι ψηφίζουμε χωριστά. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αυτή που έλειπε λοιπόν, 130 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 29, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, Επαλήθευση για την 137. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση η ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12-12. Καλά κάναμε και παληθέσαμε. Συμβαστική τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν Αλλάζουμε σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε Συμβαστική τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα, συνάδελφοι. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της συμβαστικής τροπολογίας 1. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική, α όχι, πρέπει να ψηφίσουμε. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8, επειδή κατέπεσε συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία ε, συμβαστική 13, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση. Επαλήθευση για την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται, ναι. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές καταπίπτει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18, όχι. Συμβαστική τροπολογία 9, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αφήνουμε αρκετές. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Πολύ καλή τροπολογία. Αποχές. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε, δεν πρόσεχα. Υπέρ της 29. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της 29, απλώς για να είμαστε σίγουροι. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Πρώτα η 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16. All those in against, abstentions carried. 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50, την ψηφίζουμε ξεχωριστά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Ναι, ναι. Άρχεται η ψηφοφορία για την 64. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για λίγο. Έχετε δίκιο. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 75. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεν ε, σηκώνετε πάντα τα χέρια σας και δεν καταλαβαίνουμε. 76 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. Μία παλήθευση για την 76. Πέρασε ψηφοφορία. Ναι, είναι σαφές. Εγκρίνεται. Δεν είδα το ΕΛΚ να μας λέει τι θέλει. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έχουμε τώρα την ε, γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ που καταπίπτουν όλες. Δεν έχουμε τίποτα να ψηφίσουμε λοιπόν από τη γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ. Τα πάντα καλύπτονται από άλλες τροπολογίες. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι γιατί είναι ονομαστική κλίση πέραση ψηφοφορίας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Έλλη Σλάιν, την εισηγήτρια, τους και εισηγητές, το προσωπικό. Οι συμβιβασμοί απαιτούν πολλή δουλειά, ε, αλλά έτσι διευκρινίζονται οι θέσεις μας και είναι σαφέστερες και οι ψηφοφορίες μας. Ε, όταν ακουστεί προς τα έξω καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ε, είναι σημαντικό να ψηφίσουμε τις τροπολογίες γιατί αλλιώ είναι ένα χάος τα πράγματα. Μισό λεπτό συνάδελφοι. Περιμένουμε τον κύριο Ποπόφσκι στις 6 ώρα. Θα ελέγξουμε. Μην φύγετε ακόμα. Να δούμε τι ώρα θα έρθει. Να σας εξηγήσω. Στην αρχή ήταν να έρθει η κυρία Μογκερίνη. Δεν μπορούσε να έρθει, θα έρθει κάποια άλλη συνεδρία. Θα έρθει ο κύριος Ποπόφσκι στις 6 ώρα, αλλά έχει πρόβλημα με το ταξίδι του και θα ελέγξουμε αν είναι εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική συνεδρία. ήταν μια πολύ σημαντική συνεδρία Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα και θεωρούμε ότι ήταν σημαντικό να μάθουμε τι έγινε σε αυτό το Συμβούλιο. Διακόπτουμε μέχρι τις 6 και 4 γιατί ο κύριος Ποπόφσκι μόλις προσγειώθηκε. 6 και 4 λοιπόν, σε μισή ώρα. Διάλειμμα μισή ώρα. Σας παρακαλώ να ξανάρθετε να ακούσετε τον κύριο Ποπόφσκι στις 6 και 4. Μην φύγετε, μην πιείτε πολλούς καφέδες, 6 και 4 εδώ.